Danke. Chiedo, chiedo cortesemente, please, sit down, please. Please. Buongiorno a tutti. Καλημέρα σε όλους. Κυρίως από την έναρξη της συνεδρίας της Επιτροπής μας, της διδακτικής συνεδρίας δηλαδή, και καλωσορίζω όλα τα μέλη θερμά, τα πολυάρεθμα νέα μέλη αυτής της Επιτροπής και καλωσορίσατε και εκ νέου και τα παλιότερα μέλη. Να θυμίσω σε όλους και να σας ζητήσω από όσους δεν έχετε δουλειά εδώ. Να θυμίσω σε όλους ότι στόχος αυτής της συνεδρίασης είναι η εκλογή του Πρόεδρου και των τεσσάρων αντιπρόεδρων. Οπότε δεν επιτρέπονται συζητήσεις, ερωτήσεις που δεν έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο αυτό ε, θέμα και αυτή την ημερήσια διάταξη. Η σειρά των εκλογών, όπως γνωρίζετε, είναι Πρώτα η εκλογή του Προέδρου και στη συνέχεια έχουμε εκλογή των Αντιπροέδρων Καθενό ξεχωριστά. Υπάρχουν εδώ κάποια αναπληρωματικά μέλη, αναπληρώνουν τους, τα, τακτικά μέλη που πρέπει ρητά να τους αναφέρω, γιατί όπως γνωρίζετε, για να προχωρήσουμε στις εκλογές πρέπει να έχουμε λεπτομερώς τα μέλη, τα αναπληρωματικά. Ξεκινώ από το ΕΛΚ. Λοιπόν, ο συνάδελφος Μπένστεν αντικαθίσταται από την Έστερ Ντελάγκε. Η κυρία Ντέλερ από το Βέρνερ Λάγκεν. ναι, που αξίζει μια ένα χειροκρότημα. Η κυρία Άγγελα Νίμπλερ αντικαθίσταται από τον Μάρκος Πίμπερ. Ο κύριος Ματριτσέλο από τον συνάδελφο Σαβίνη. Σαοντάργας από ε, ε, Εστέμπαν Γκονζάλες Πόνς και από τους σοσιαλιστές Μπαλτσίτης αντικαθίσταται από τον κύριο Μάνκα. Στανισέβης από τον Γιακόφα. Γκίρεκ, Άνταμ Γκίρεκ αντικαθίσταται από τον Όλε Λούντβικσον. Νταν Νίκα από το Σόριν Μόιζα. Από το ECR. Ο συνάδελφος Γκορμπάρτσιτς, ελπίζω να μην το σκότωσα το όνομά του, από το Σαν Ποτέρο από την Άλντε, η Άγγελα Μπλίναρ από τον Πάβελ Τελίκα. Από τους Πρασίνους, ο Μπούτι Κόφερ αντικαθίσταται από τον Γιάννη Ξαντό. και ολοκληρώνω από την ε, EFT ο Μπορέλη από τη Λάουρα Φεράρα. Παρακαλώ. Α, εντάξει, λάθος. Είναι παρόν, είναι παρόν. Ωραία. Πρόκειται για αντικαθιστάτες λοιπόν που ε, προβλέπονται από τη γραμματεία. Όπως ξέρετε δεν γίνεται να κάνει κανείς αντικατάσταση παρά μόνο πριν την ψηφοφορία και έτσι τώρα έχουμε ολοκληρώσει και το θέμα των αναπληρωματικών μελών. Όσοι ανέφερα μπορούν να ψηφίσουν σήμερα. Ε, ζητώ λοιπόν τώρα από τη γραμματεία, αν έχουμε απαρτία, μάλιστα, Ξέρετε ότι η απαρτία για τη δική μας επιτροπή είναι 17 μέλη, αλλά φυσικά είμαστε πολύ περισσότεροι σήμερα παρόντες και προχωράμε τώρα, αφού έχουμε λοιπόν απαρτία, στην εκλογή του Προέδρου. Θα ρωτήσω εάν υπάρχουν υποψηφιότητες. Κύριε Κάριτς, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Εξ ονόματος του ΕΛΚ θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Γέρζη Μπούζεκ ως πρόεδρο της Επιτροπής αυτής. Ακούσατε λοιπόν, ε, υποψήφιος είναι ο συνάδελφος Μπούζεκ και θέλω να το ρωτήσω αν δέχεται την υποψηφιότητα. Μάλιστα, το δέχομαι. Είμαι υποψήφιος. Ναι. Ε, δεν πρόλαβα να ρωτήσω αν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Όχι. Οπότε, να προτείνω, αν θέλετε, να προχωρήσουμε διαβοή στην εκλογή του κυρίου Μπούζεκ ως Προέδρου της Επιτροπής. con questo applauso di acclamazione eh, il Ωραία λοιπόν, ο κύριος Πρόεδρος του, πρώην Πρόεδρος του Κοινοβούλιου είναι τώρα Πρόεδρος αυτής της Επιτροπής, συγχαρητήρια. Δεν έχω παρά να σας παραδώσω αυτή τη θέση και σας εύχομαι καλή δουλειά σε αυτή την Επιτροπή. Uh, thank Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου. Για το ότι εμπιστευτήκατε λοιπόν εμένα και θέλω να σας πω ότι θα είμαι ανοιχτός, δίκαιος. Έχουμε τον εσωτερικό μας κανονισμό, τον οποίο θα τηρώ και βέβαια είναι και πολύ σημαντικό εργαλείο σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ας πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της μερισιάς διάταξης, δηλαδή στην εκλογή των τεσσάρων αντιπροέδρων. Δεν θα τους εκλέξουμε μαζί, έναν έναν, ξεχωριστά. that... Θα ήθελα να σας πω βέβαια ότι τα αναπληρωματικά ε, μέλη που αντικαθιστούν κάποιο τακτικό μέλος φυσικά ψηφίζουν. Σας είπε τα ονόματα κυρία Τόγια πριν από λίγο, πριν ξεκινή, όταν ξεκινήσαμε τη συνεδρίασή μας. Απλά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μπορεί να χρειαστούμε κανένα 20 λεπτό, μέχρι να ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία. Ίσως υπάρχουν αλλαγές, προτείνεται κάποια αλλαγή. Εάν ναι, πριν ανακοινώσω ότι προχωράμε σε ψηφοφορία παρακαλώ, να μας γνωστοποιήσετε τις αλλαγές. Λοιπόν, όπως είπαμε έχουμε απαρτία, περνάμε λοιπόν στην εκλογή καταρχάς του ή της πρώτης ή πρώτου πρόεδρου Υποψηφιότητες παρακαλώ. Κυρία μου, σας ακούμε. Ε, ναι, κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα την Πατρίσια Τόγια, την καλή συνάδελφο, να την προτείνουμε για τη θέση της πρώτης αντιπρόεδρου. Πρόεδρος. Εκ μέρους της ομάδας σοσιαλιστών δημοκρατών, έτσι μάλιστα, ωραία. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Τόγια, να σας ρωτήσω. Καταρχάς, συμφωνείτε με την υποψηφιότητα, δέχεστε, δέχομαι. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Επόμενη ερώτηση προς την κυρία Τόγια. Ή μάλλον υπάρχουν άλλοι υποψήφοι, καταρχάς. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος άλλος υποψήφιος. Προτείνω λοιπόν κάτι πολύ απλό, διαβοής, να εγκρίνουμε την υποψηφιότητα. Κυρία Τόγια, αγαπητή Πατρίτσια, συγχαρητήρια. Σε προσκαλώ να έλθεις να καθίσεις εδώ, στο Προεδρείο, δίπλα μας. Left few Πριν από λίγο έφυγες από τη θέση σου, ε, ξαναέλα τώρα. Στην πολύ σημαντική θέση πλέον της πρώτης αντιπροέδρου. Περνάμε λοιπόν τώρα στην εκλογή του δευτέρου αντιπροέδρου της Επιτροπής μας. Ερωτώ, υποψηφιότητες υπάρχουν. Βλέπω εκπρόσωπο από την ομάδα ECR. Παρακαλώ, να συστηθείτε κιόλας. Ευχαριστώ. Ashley Fox είναι το όνομά μου αντικαθιστώ τον ε, Charles Chichester, μεγάλη τιμή για μένα, ήταν ένας καλός συνάδελφος και με μεγάλη χαρά θα ήθελα να προτείνω έναν άλλο καλό συνάδελφο, τον καθηγητή Χένκελ, για τη θέση του δεύτερου του Προέδρου. My question is, as Όπως και πριν, λέει ο Πρόεδρος, ερωτώ. Καταρχάς, υπάρχουν άλλες υποψηφιότητε. Δεν βλέπω κάποιον να προτείνει κάποιον άλλον. Α, βέβαια, πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Χέγκελ αν συμφωνεί. Δέχεστε να είστε υποψήφιο. Δέχομαι. Σα ευχαριστώ πολύ, πρόεδρος. Διαβοής παρακαλώ, όπω και πριν να εκλέξουμε τον δεύτερο μα αντιπρόεδρο. Σα ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφε, σα συγχαίρω και σα καλώ να έλθετε να καθίσετε εδώ στο Προεδρείο μαζί μα. Well, as usual, in each committee very quickly. Fantastic. Πολύ γρήγορα πηγαίνουμε. Φανταστικά. Έχουμε και πολλά να κάνουμε στη νέα αυτή κοινοβουλευτική περίοδο και καλό είναι να οργανωθούμε έτσι γρήγορα γρήγορα. Everybody the same way. Good. Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε στην εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου. Παρακαλώ, προτάσεις. Από ό,τι βλέπω η Γκου έχει να κάνει μια πρόταση. Αγαπητέ συνάδελφοι. Μου είναι ο Κλής Εκ μέρου τη Ενωμένη Αριστερά και Βόρεια Πράσινη Αριστερά προτείνω τον ε, συνάδελφο Μυροσλάβ Ράνστοφ για τρίτον αντιπρόεδρο. Μυροσλάβ Ράνστοφ. Μιστέρ Ransdorf. Θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Ράνστοφ να μας πει αν συμφωνεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με την πρόταση. Other proposals. Υπάρχουν άλλες προτάσεις, άλλες υποψηφιότητες, συνάδελφοι. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, επομένως... Διαβοής να εκλέξουμε τον τρίτο μας αντιπρόεδρο. Τέλεια. Αγαπητέ συνάδελφοι, σας συγχαίρω. Αγαπητέ Μύροσλαβ, έλα να καθίσεις και εσύ μαζί μας στο Προεδρείο. Ε... Last but not least. Τέλος, εξίσου σημαντικό όμως, εκλογή του τέταρτου αντιπρόεδρου. Candidates. Mrs. Ferreira. Υποψηφιότητες παρακαλώ. Uh, Madame Ferreira. Κυρία Φερέρα. Ή Φεράρα. Φεράρα, ομάδα EFTD. Καλησπέρα Πρόεδρε. Εξ ονόματος ε, της ομάδας EFTD θα ήθελα να θέσω υποψήφιο τον κύριο Ταμπουράνο για την τέταρτη ε, αντιπροεδρία της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ντάριο Ταμπουράνο, δέχεστε την υποψηφιότητα αυτή. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν, το δέχεστε. Αλλά βλέπω και άλλη μια υποψηφιότητα. Εξ ονόματος του Άλντε. Έχουμε τον κύριο Φέντερικ Φέντερλε που ζητά το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, δεν είμαι εγώ υποψήφιος, αλλά εξ ονόματος της Άλντε θα ήθελα να υποβάλω μια υποψηφιότητα που είναι ο κύριος Πέτερσεν από την Σουηδία. Μάλιστα. Κύριος Μόρτεν Πέτερσεν λοιπόν είναι υποψήφιος. Κύριε Πέτερσεν, δέχεστε την υποψηφιότητα? Μάλιστα τη δέχομαι. So we have uh, two candidates in the case... Μάλιστα έχουμε δύο υποψηφίους. Λοιπόν, στην, υπόθεση, περίπτωση δύο υποψηφίων προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία θα γίνει. Και να σας δώσω κάποιες πληροφορίες που είναι πολύ σημαντικές τώρα στην αρχή. Βεβαίως Κάθε μέλος που συμμετέχει στην ψηφοφορία έχει μία ε, ψήφο. Στον πρώτο γύρο Για να εκλεγεί ο υποψήφιος θα πρέπει να ε, έχει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Εάν δεν επιτευχθεί αυτό στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο θα έχουμε πλειοψηφία των ψηφισάντων. Εάν υπάρξει ισοψηφία, τότε ο γυρεότερος των υποψηφίων εκλέγεται. Νομίζω πως αυτά είναι όλα σαφή. Έχει κάποιος ερώτηση? Μάλιστα, παρακαλώ. Ονομάζομαι Πίτρ Έριξον, είμαι από τους Πράσινους. Θα ήθελα να έχω μια εξήγηση από την άλλη, γιατί υποβάλλουν άλλον υποψήφιο, αφού έχουν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις μεταξύ μας στην... για τη συμπροεδρία. Είναι δυνατόν να εξηγήσετε στην Επιτροπή μας, αλλά είναι, υπάρχει ελευθερία Κάθε πολιτική ομάδα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Όπω γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο αγαπητό συνάδελφο Έριξον, οι πλειοψηφίε σχηματίζονται από συναμαχίε, συνασπισμού. Εκτό εάν ένα μόνο κόμμα έχει την απόλυτη πλειοψηφία, πράγμα που δεν συμβαίνει. Είναι δημοκρατικό μα δικαίωμα να υποβάλουμε υποψηφιότητα ω πολιτική ομάδα. Μάλιστα. Καταλάβαμε αυτή την εξήγηση. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Να μην σας ε, ενοχλήσω κιόλας, αν θέλετε, να θέσετε κι άλλες υποψηφιότητες. Λοιπόν, δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη υποψηφιότητα. Λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα ψηφίσουμε με μυστική ψηφοφορία και με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Οπότε χρειάζεστε τις κάρτες σας. Κάποιος δεν έχει κάρτα. Κύριε Πρόεδρε, ήμουν στην προηγούμενη συνεδρίαση εδώ, στη συνεδρίαση ίντα και είχα αφήσει την κάρτα μου εδώ στη σχισμή, όμως όταν ήρθα οι υπηρεσίες είχαν αφαιρέσει την κάρτα. Μήπως κάποιος άλλος είναι χωρίς κάρτα ψηφοφορίας, γιατί μπορούμε να σας δώσουμε μια κάρτα αντικατάστασης σε λίγα λεπτά. Είναι κάποιος άλλος που δεν έχει κάρτα? It will take us maybe to minutes. Τρία με πέντε λεπτά. Is original. Ωραία, έχετε λοιπόν την πρωτότυπη σας κάρτα, ούτε καν αντικατάσταση. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στο, στο προσωπικό μας, αγαπητοί φίλοι. Άλλος κανείς λοιπόν με ερωτήσεις. Ωραία. Τώρα, στρέφομαι στον κανονισμό. Ε, Έχουμε λοιπόν δύο υποψηφιότητες, γνωρίζουμε τα ονόματα, Πέτερσεν και Ταμπουράνο. Τα δύο αυτά πρόσωπα έχουν κατέλθει υποψήφιοι. Εγώ, όπως είδατε, τα ανέφερα αλφαβητικά. Θα σας παρακαλέσω να τηρείτε αυτή η αλφαβητική σειρά. Πέτερσεν, Ταμπουράνο. Αυτούς έχω στην λίστα. Τώρα αν αρχίσουμε την ψηφοφορία, θα πω αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is open. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει. Και να θυμηθείτε ότι το πράσινο κουμπί αντιστοιχεί στον πρώτο υποψήφιο. Το κόκκινο στον δεύτερο. Δηλαδή, Πράσινο κουμπί σημαίνει ότι ψηφίζετε υπέρ του κυρίου Πέτερσεν, κόκκινο κουμπί σημαίνει ότι ψηφίζετε υπέρ του κυρίου Ταμπουράνο. Ψηφίζετε τον ένα υποψήφιο, αν θέλετε να ψηφίσετε τον κύριο Πέτερσεν, πατάτε το πράσινο κουμπί. Αν θέλετε να ψηφίσετε τον κύριο Ταμπουράνο, το κόκκινο. Αυτό είναι όλο που έχετε να κάνετε. Εμείς θα καταμετρήσουμε όλες τις ψήφους ηλεκτρονικά. Όπως είπα η ψηφοφορία είναι μυστική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εάν κάνετε λάθος, όσο δεν έχω κλείσει την ψηφοφορία, μπορείτε να αλλάξετε, να αντιπράσινο το κόκκινο ή αντί το πράσινο. Κανένα προνόμιο για οποιονδήποτε. Όταν πω έληξη ψηφοφορία, the vote is closed, σημαίνει ότι πια δεν αλλάζει τίποτα. Θα έχουν καταχωριστεί οι ψήφοι σας. Θα κάνουμε πρώτα μια δοκιμαστική ψηφοφορία, που σημαίνει ας πούμε τι να ψηφίσουμε. Υπέρ Βραζιλίας ή υπέρ Αργεντινής, ας πούμε, έτσι, για το ποδόσφαιρο, ναι. Βραζιλία ή Αργεντινή. Ας πούμε, Βραζιλία. Α, έχει ανατρέψει ο πρόεδρος στην αλφαβητική σειρά, μου αρχίσει από τη Βραζιλία. Α, αλφαβητική σειρά. Ναι, σωστά. Λοιπόν, Αργεντινή πράσινο και Βραζιλία κόκκινο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Ψηφίσατε. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Τέλος, έληξη η ψηφοφορία. Ας δούμε τώρα. Νομίζουμε ότι τα έχει, τα έχει αντιστρέψει ο Πρόεδρος, πάντως είναι ψήφοι 31 και 22 υπέρ ε, Αργεντινής και Βραζιλίας. Και τέσσερις που δεν αναποφάσιστη ας πούμε έτσι. Τώρα, στο πρώτο γύρο, χρειαζόμαστε απόλυτη πλειοψηφία για να είναι θετικό το αποτέλεσμα. Στον δεύτερο γύρο, ο μεγαλύτερος αριθμός ψήφων, γιατί έχουμε δύο υποψηφίους θα είναι αυτό που θα ισχύσει. Συμφωνεί. Και τώρα ας αρχίσουμε. Ε, έχετε κατανοήσει καλά τη διαδικασία. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Έληξε η ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα έχει ως εξής. 37 ψήφοι υπέρ του κυρίου Πέτερσεν. 22 λέει ο πρόεδρος υπέρ του κυρίου Ταμβουράνο. Επιτεύθηκε η, απόλυτη πλειοψηφία υπέρ του κυρίου Πέτερσεν. Και συγχαρητήρια και Πέτερσεν. Σας παρακαλώ αγαπητέ συνάδελφε, συγχαρητήρια πρώτα και ελάτε να καθίσετε δίπλα μας. Okay. 17, yes, 17, sorry. Συγχωρείτε, το αποτέλεσμα είναι 17 διορθώνει η πρόεδρος. Έτσι, 37-17. Πάντως επιτέθηκε η πλειοψηφία. Έχω και ορισμένες ανακοινώσεις ε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν από το τέλος της συνεδριάσεώς μας βλέπετε εδώ το Προεδρείο μας, το Προεδρείο της Επιτροπής μας. Μύροσλαβ, να σφίξω το χέρι σας. Λοιπόν, ορισμένες ανακοινώσεις που ίσως αποδειχθούν σημαντικές για όλους σας. Ορίστε, παρακαλώ, υπάρχει μια ερώτηση. Το... Εγώ ήθελα απλά να κάνω μια δήλωση γιατί εδώ βλέπουμε σήμερα σε όλες τις επιτροπές μια παραβίαση της μεθόδου DON'T που αποδεικνύει πως αυτό το πρότυπο για την Ευρώπη δεν επιτρέπει ούτε τη θεμητή επίκριση. Οι μειοψηφίε αποκλείονται από τα καθήκοντα των θεσμικών οργάνων. Μιλάμε και για το κίνημα των πέντε αστεριών που ωστόσο συγκέντρωσε μεγάλη πλειοψηφία των Ιταλών ψηφοφόρων. Το να καταγγέλουμε τις δημοκρατικές, τις, μάλλον τις λανθασμένες πρακτικές δεν σημαίνει πως δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα και με, με τιμά του ότι είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής που θεωρώ ότι είναι στρατηγική σημασία για τις μελλοντικέ ε, γενναίες. Αυτή μου η προσήλωση θα είναι καθοριστική για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας, ενώπιον της Ευρώπης και ελπίζω πως το πρότυπο της Ευρώπης που θα οικοδομήσουμε από κοινού θα είναι υποδειγματικό παρά τα όσα συμβαίνουν σήμερα για ειρήνη, πραγματική δημοκρατία, συμμετοχή και ευημερία για όλο το ε, σφαιρικό αποτέλεσμα για τον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ. Uh, well, let me warmly welcome once again. Σας συγχαίρω πάντως όλες και όλους που εξελέγετε. Συγχαίρω και όλα τα νέα, τα νεοσυρχόμενα μέλη. Είμαστε μια μεγάλη επιτροπή, η τρίτη μεγαλύτερη, τρίτη κατά μέγεθος δηλαδή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρύτατο περιεχόμενο του χαρτοφυλακίου μας. Έχουμε πολλά θέματα, ε, βιομηχανία, μικρές και μεσές επιχειρήσεις, έρευνα, καινοτομία, ψηφιακή οικονομία, ψηφιακή ατζέντα και βεβαίως την ενέργεια. Πολύ σημαντική υπόθεση και σημαντικός κλάδος. αυτά που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες εβδομάδες είναι πρώτα η έγκριση των υποψηφίων επιτρόπων μετά από τις θερινές διακοπές. Στην επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα προβούμε σε ακρόαση του κυρίου Φερότσι που είναι υποψήφιος επίτροπος εις αντικατάσταση του κυρίου Ταγιάννη. Οι κύριοι Ταγιάννη και Λεβαντόφσκι είναι τώρα ευρωβουλευτές. Έχουμε μεταξύ μας και πρώην υπουργούς και επιτρόπους, αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλοι σας είστε επαγγελματίες υψηλωτά του επίπεδου. Το γνωρίζουμε από τα βιογραφικά σας σημειώματα. Συναπαρτίζεται λοιπόν μια πολύ σημαντική κοινοβουλευτική επιτροπή. Άλλο δεύτερο σημαντικό θέμα, 22 Εβδόμου, θα συζητήσουμε τη στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας που ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ζητήσω και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας ενημερώσουν για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων της συμφωνίας με τις Ενωμένες Πολιτείες, TTIP. Και θα έχουμε, όπως είπα, όλα αυτά τα σημαντικά θέματα, τιμές της ενέργειας, το κλίμα βεβαίως, την ψηφιοποίηση και την ηλεκτρονική αγορά, την, την εκ νέου εκβιομηχάνηση περιοχών. Όλα αυτά είναι στην ατζέντα μας για μέχρι τέλος του χρόνου, με, πάνω στην κοινοβουλευτική μας περίοδο. Ευχαρίστω να συνεργαστώ μαζί σας, με τους συντονιστές, αλλά και με κάθε μεμονωμένο μέλος. Είμαι βέβαιος ότι με κοινή προσπάθεια μπορούμε να επιτύχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε πέντε χρόνια μπροστά μας. Καλή επιτυχία λοιπόν εύχομαι σε όλες και όλους εσάς και εμένα. Ευχαριστώ.